ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτό το πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Πέρα στη συζητήσεω, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Πηγαίνουμε στο επόμενο σημείο της ημέρησιας διάταξης της απογευματινής. Κοινή συζήτηση. Αυτή αφορά το Μητρό Διαφάνειας. Η πρώτη έκθεση είναι του κυρίου Κασίνη και αφορά τη Διοργανική Συμφωνία σχετικά με ένα κοινό μητρό διαφάνειας και μετά έχουμε τη δεύτερη έκθεση που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού σε συνέχεια της δημιουργίας κοινού μητρώου διαφάνειας. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ο κύριος Κασίνη, που είναι ο εισηγήτης μας, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρία, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μία εισήγηση θα κάνω και για τα δύο θέματα γιατί αφορούν το ίδιο. Με αυτή την ψηφοφορία και την ακολουθούσα ψηφοφορία ολοκληρώνεται μια πεδίο διαπραγματεύσεων των ομάδων εργασία, τη οποία προέδρευσε η πρόεδρο κυρία Βόλη, μαζί με του συναδέλφου όλων των πολιτικών ομάδων με την αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, υπό τον Επίτροπο Σεύκοβιτ, που οδήγησε στη σύνταξη ενό κειμένου για τη συμφωνία μεταξύ θεσμικών οργάνων για ένα κοινό μητρό διαφάνεια. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ σε μερικού μήνε μετά την σύνταξη της εκθέσεως ε, τίμασε και κάποιο κείμενο που αφορά του διάφορου τροποποίησεις του κανονισμού. Εγώ εξεπλάγει τα μάλα λόγω της προσοχής που έδωσε η κοινή γνώμη σε αυτή τη συμφωνία για το Μητρό Διαφάνειας. Φοβούμε ότι ίσως να περιμένουν αποτελέσματα μεγαλύτερα από, από τα επιδιωκόμενα. Διαφάνεια ε, είναι και η προάσπιση της σωστής πολιτικής δράσεως αλλά δεν είναι ένα όργανο που πλήττει τη διαφθορά στο επίκεντρο. Τα διάφορα επεισόδια που είδαμε ότι κάποιοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να διαφύρουν κάποιους βουλευτές ε, βγαίνουν και εκτός ανέα από το Κοινοβούλιο. Και εκείνοι που διαφύρουν ξέρουν πώς να το κάνουν για το, ώστε να μην είναι εντοπίσιμοι και τα, να μην διαπιστώνουν την ταυτότητά τους. Λοιπόν, το μέσο το δέον είναι ο ποινικό κώδικας. Και, και αν δεν αρκεί σε επίπεδο 100 μελών, θα αρκεί να διαβάσετε τα άρθρα από 82-86 της συνθήκης Λισαβόνας που αντικατοπτρίζουν κατά πόσο στη διαφθορά των Ευρωπαίων βουλευτών μπορούν να, δώσουν, να θεωρηθούν σαν ένα δίκημα διασυνοριακό ή κάτι που στέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας και αν χρειάζεται να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ενότητα. Το μητρό της διαφάνειας έχει πιο μετριοπαθή στόχο. Σε κάποιες χώρες ο όρος του λόμπιστ έχει αρνητική χρειά. Σε άλλες χώρες η δραστηριότητα των ομάδων πίεσης λόμπι θεωρείται σχεδόν ε, δημόσιο έργο. Διότι ε, ε, προωθεί και κάποια προβλήματα που ήταν άγνωστα χωρίς τα λόμπι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό, διότι πολύ συχνά τα θέματα που, αντιμετωπίζουν ε, οι βουλευτές είναι αρκετά περίπλοκα και τεχνικής φύσης. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ ε, διαφόρων, συμφερόντων. Οι, λόμπι, ε, τα, οι λομπίστες είναι χρήσιμοι σε αυτή την περίπτωση, προωθούν διάφορα συμφέροντα, έτσι πρέπει να θεωρούνται. Μπορεί να αντίθετα τα συμφέροντα. Εγώ ήμουν δικαστής και μπορώ να πω ότι η αντίφαση μεταξύ των αντιθέτων μέρων ίσως είναι ένας τρόπος να βρει κανείς τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Ε, λοιπόν, λομπίστε ή μεταφορεί συμφερόντων που ακολουθούν. Όμω όμως ο δικαστής θα πρέπει να είναι εξάρτητος, να έχει ελευθερία σκέψη όπως ο δικαστής και να κινείται προ το κοινό όφελο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε, θεσπίστηκε αυτό το μητρό διαφάνεια κοινή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου. Και ελπίζουμε και το Συμβούλιο σύμφωνα, ε, σύντομα να συμφωνήσει. Ε, λοιπόν, θα, θέλουμε να προστατεύσουμε, να δημιουργήσουμε ένα μητρό όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία που εντοπίζουν την νομική δομή και η οικονομική δομή εκείνου που θέλει να κινείται σε αυτό το χώρο. Το δημόσιο μητρό συμπεριλαμβάνει και διάφορους φορείς που θέλουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικής, ευρωπαϊκής, κόμματα, περιφέρειες, εκκλησίες μπορούν να ε, συμμετέχουν ε, και θα πηγαίνουν στο ε, Μητρό μόνο αν υπάρχει συγκεκριμένο γραφείο αυτών που κινείται εντό Ευρωπαϊκή Ενώσης. Τότε μπαίνει στο Μητρό. Διαφορετικά έχουμε άλλο καθεστώς των άλλων φορέων. Πρέπει να τροποποιηθεί και ο κανονισμό για το Μητρό. Το είπαμε αυτό. Έχουμε δύο εκθέσει. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό για μεγαλύτερη, πληρέστερη διαφάνεια. Μετά από προβληματισμό θα σπιστούν και άλλοι κανόνες. Ο αριθμός, στο άρθρο 9 αναφέρεται η δυνατότητα να αναφέρονται τα διάφορα στοιχεία. Χρειάζεται μεγάλο άνοιγμα για δυνατότητα αναθεώρηση. Οι τροποποίησει που θέλουν να θέσουν δεσμεύσει κλείνουν την προσέγγιση. Εάν μετάσχει και το Συμβούλιο στη Συμφωνία θα υπάρξει μεγάλη συνένεση και στο Κοινοβούλιο. Χρειάζεται δράση και διαφάνεια. Και ελπίζω τελικά να υποστηριχθούν αυτά τα μέτρα που προτείνονται μέσω της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ κύριε Κασίνη. Στρέφομαι τώρα προς την Υπουργό, την κυρία Γιώρη που θα εκφραστεί εκ μέρους της ε, Προεδρίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τις ε, απόψεις του Συμβουλίου ε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική για την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και ιδίως των ε, ευρωπαϊκών, διότι όπως το γνωρίζετε λέγεται ότι οι ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν απομακρυνθεί από τους πολίτες και δεν είναι διάφανα. Ενώ πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των συναλλαγών και προς τα έξω. Και όταν οι πολίτες έρχονται και στρέφονται σε εμά για να λύσουμε τα προβλήματά τους απαιτούν υψηλές προϋποθέσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό διαφανεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζω την πρόταση του κυρίου Κασίνη και αν ψηφιστεί η έκθεση αυτή θα αποτελέσει βάση για διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρξει ένα κοινό μητρό και να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη και με πράξεις εις την ανάληψη αυτών των ευθυνών. Βεβαίως γνωρίζω ότι το Συμβούλιο έχει προσεγγιστεί τελευταίως για να συμμετάσχει κατά κάποιον τρόπο στο Μητρό Διαφανείας ενώ δεν θα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία διότι το Συμβούλιο λόγω της φύσεώς τους δεν επηρεάζεται από τα λόμπι. Τα λόμπι δεν έρχονται στο Συμβούλιο σαν ευρωπαϊκό θεσμό αλλά στα κράτη-μέλη για να κάνουν τη δουλειά τους. Παρόλα αυτά το Συμβούλιο είναι έτοιμο να δεχθεί ορισμένους, ε, ορισμένα μέτρα σχετικά με το Μητρό αυτό και να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να συμμετάσχουμε και εμείς στο Μητρό αυτό χωρίς όμως να πρέπει να καθυστερήσουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ των δύο εμπλεκομένων δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Αυτή στιγμή ε, εξετάζεται ένα σχέδιο πολιτικής δηλώσεως που θα ακολουθήσει τη δημοσίευση του, της προτάσεως του Μητρώου. Ευχαριστώ, δίνω το λόγο ή στον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Ε, ε, θα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό θέμα και ε, ενδιαφέρει όλους τους πολίτες για να νομιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χαίρομαι ότι υπάρχουν πέραν των 300 ήδη εγγραφών εις το μητρό αυτό το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών. Θα ήθελα να επενέσω την επικοδομητική εργασία όλων και αναφέρομαι εδώ στην κυρία Γόλης που προεδρεύει σήμερα, στον κύριο Κασίνη, τον κύριο Λάινεν και την κυρία Ντουρόν. Ήταν μεγάλη χαρά μου να συνεργαστώ μαζί σας και η εργασία αυτή είναι πολύ ισοσκελισμένη. Γι' αυτό όμως θα θα έπρεπε να υπάρξει μια πιο θετική αντιμετώπιση. Στον αφορά τη δρομολόγηση αυτού του Μητρού και θα πρέπει αυτό να γίνει τον Ιούνιο. Αυτό σίγουρα θα στείλει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θα δείχνει την αποφασιστικότητά μας για να, για να εφαρμόσουμε ε, πρακτικέ διαφανεί και σωστέ στο προσκήνιο του ευρωπαϊκό. Το Μητρό έχει σαν στόχο να δώσει στου πολίτε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την διοργάνωση των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι ασχολούνται με διαμόρφωση πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εκφράστηκαν κάποιε ανησυχίε όσον αφορά τι περιφερειακού τοπικού φορεί. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρό. Και εγώ νομίζω ότι αν διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο είναι αρκετά σαφέ ότι αυτό δεν αντικατοπτεί στην πραγματική του ταυτότητα ούτε το γεγονό ότι εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση των πολιτών κάτι που, δια, δημιουργεί το δικό του συνταγματικό σύστημα. Διαβάζοντα προσεκτικά τη συμφωνία θα διασκεδαστούν οι ανησυχίες σας. Πραγματικά το κείμενο ρητά αναφέρει ότι οι τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές δεν αναμένεται να ε, καταχωρηθούν. Και αυτό ενισχύεται και το παράρτημα 1, όπου εκεί αναφέρεται ότι οι δημόσιε αρχέ αυτέ καθ' αυτέ δεν αναμένεται να καταχωρηθούν. Οι υπηρεσίε που αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα ε, τη ε, της δεν θα συμπεριλαμβάνονται όπως προανέφερα. Και έτσι διασκεδάζονται ανησυχίε όσον αφορά το Μητρό. Τέλος, όσον αφορά τη διοργανική διάσταση. Όλοι μοιραζόμαστε την άποψη ότι επίτευγμα της κοινή μα συνεργασίας μεταξύ δηλαδή Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου θα είναι κάτι που παγιωθεί περαιτέρω με την εμπλοκή του Συμβουλίου. Και ευχαριστώ ολόθερμα την Ουγγρική Προεδρία που αλλάζει την ατμόσφαιρα στο Συμβούλιο και τελικά το Συμβούλιο θα είναι πιο θετικό και θα διερευνηθούν τρόποι για καλύτερη διευθέτηση σχέσεων Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό ε, όσον αφορά τη διαχείριση του Μητρώου. Νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα ότι τα τρία θεσμικά όργανα παίρνουν δουλειά σα σοβαρά θα βγει προς τα έξω. Ότι αντιμετωπίσουν το θέμα της διαφάνειας μαζί τα τρία θεσμικά όργανα θα είναι ισχυρό μήνυμα. Και μια τέτοια πολιτική υποστήριξη και από τα τρία θεσμικά όργανα ε, θα είναι κάτι που θα βοηθήσει στο να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τον επικοδομητικό σας ρόλο στη συζήτησή μας. Πάμε στους αγορητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Καταρχάς ο κ. Βέμπερ εκ μέρου του ΕΛΚ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, η, η, η αφάνεια είναι η βάση της δημοκρατίας και από όταν ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερη ισχύ γι' αυτό και ε, πρέπει να εξετάζουμε πάντοτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και να τον αμφισβητούμε και γι' αυτό το Μητρό Διαφανείας είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πρέπει να τονίσω ότι είναι καλό διότι για την τοπική αυτοδιοίκηση θα υπάρξουν επίσης τις ε, σαφείς ρυθμίσεις που θα τονίζουν το ρόλο τους. Θέλω να πω ότι τα, τα λόμπι δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό. Χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες για τη δουλειά μας και εμείς ε, σαν, ε, κοινο, σαν βουλευτές πρέπει να μπορούμε μετά να κινηθούμε ελεύθερα και να είμαστε περήφανοι διότι αν συγκρίνουμε με το εθνικό επίπεδο πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν λίγες χώρες στην Ευρώπη που έχουν τέτοιο μητρό διαφανείας στο Βερολίνο στη χώρα μου δεν υπάρχει τέτοιο μητρό διαφανείας και άρα εμείς έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ίσως στο Συμβούλιο δεν χρειάζεται διότι υπάρχει υπάρχει λιγότερη επέμβαση των λόμπι, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να προσχωρήσει και το Συμβούλιο στο Μητρό και σαν κοινοβουλευτική ή στο μέλλον εάν θέλουμε να εργαστούμε χωρίς να μας επηρεάζουν τα λόμπι, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους συνεργάτες μας να επανδρωθούμε καλύτερα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριο Γκρότη για δύο λεφτά εν ονόματι των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον εισηγητή και για όλους τους συμμετέχοντες διότι σήμερα ή μάλλον αύριο μετά την ψηφοφορία θα στεφθεί ε, μία μακριά πορεία εργασίας και θα είναι μία ωραία μέρα για την Ευρώπη, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επέτρεψε να καταρτήσουμε ένα μητρό διαφανείας. Είναι ένα σταθμό ο οποίος χρήζει, βοήθει, χρήζει επίσης. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό το μητρό αυτό. Πρέπει να λεχθεί εδώ σαφώς. Και ε, όπως ε, ελέγχθη από τον ε, Επίτροπο υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή όμως θα συμβάλλει σε αυτή την τροποποίηση κατά τρόπον ώστε το μητρό στο μέλλον να γίνει υποχρεωτικό. Και ε, από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι είναι δύσκολο κάτι τέτοιο αλλά θα ήθελα να προσχωρήσει και το Συμβούλιο διότι τότε θα είναι ε, πλήρες το Μητρό εάν εκπροσωπούνται από κοινού και ε, τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ένα Μητρό που είναι υποχρεωτικό και γι' αυτό θα δεχθούμε μία τροπολογία μίας άλλης πολιτικής ομάδας ότι τα ποσά τα οποία αναφέρονται εις το Μητρό Διαφανείας για εργασία λόμπι θα πρέπει να καταγράφονται ε, και γι' αυτό ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν στη διατύπωση των ε, τροπολογιών συμβιβαστικά για να φύγει η μαύρη αυτή κοιλίδα που δημιούργησαν τα λόμπι εδώ. Ο κύριος Ντάφ για δύο λεπτά εν ονόματι της, φιλελεύθερης, ε, ομάδας των φιλελευθέρων. Oh, uh, uh, Τα πρόσφατα σκάνδαλα εξέθεσαν την ε, εξουσία δεδομένου ότι είναι μεγάλη η επιρροή που μπορούν να έχουν ε, οι εκπρόσωποι των λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι φιλελεύθεροι χαιρετίζουν τη δημιουργία αυτού του ε, μητρώου διαφάνειας το οποίο παρά το γεγονός ότι είναι προαιρετικό θα μπορέσει να προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια κύριες υπέρ της παραγράφου 9 της έκθεσης που αφορά τη διαφάνεια που καλεί το Προεδρείο να δημιουργήσει ένα σύστημα νομοθετικού αποτυπώματος όπου οι εισηγητές θα μπορούν να καταγράφουν τα μητρώα για τα οποία έχουν δεχθεί προσώπους των λόμπι πριν να νομοθετήσουν. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα βήμα προς τα μπρος για τη βελτίωση της νομιμότητας του Κοινοβουλίου και της ποιότητας των νομοθετικών μας πράξεων. Το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αν το Συμβούλιο δεν συμμετάσχει στην όλη διαδικασία, αλλά χαιρετίζω τα διάφορα βήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι διατεθειμένο να κάνει, διατεθειμένο να κάνει το Συμβούλιο και ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία για τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το απόγευμα. Κύριε Ντάφ, από τον κύριο Γκρότα έχετε μπλε κάρτα. Ευχαριστώ. Ε, σχετικά με το νομοθετικό αποτύπωμα. Πιστεύετε ότι ένα νομοθετικό αποτύπωμα και πρέπει να καθορίσουμε ακόμη την έκτασή του ε, θα μπορέσει να περιορίσει την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς εσείς ε, βλέπετε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το νομοθετικό αποτύπωμα θα μπορέσει να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι όλες ε, οι προσπάθειες, αν ε, είναι επιτυχείς, θα οδηγήσουν σε μια ευρύτερη χρήση. Αλλά θα έπρεπε να περιοριστεί εις τους εισηγητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ε, έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, διατύπωση και ε, για να να δημοσιεύσουν ε, τις συζητήσεις που είχαν σε επίσημες συνεδριάσεις και το αποτέλεσμα των εργασιών τους κατά τρόπον ώστε να υπάρξει ε, ένα αποτελεσματικό σύστημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους εμπειρογνώμονες και τους επαγγελματίες εκτός του Κοινοβουλίου για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη σύνταξη των εισηγήσεων. Ευχαριστώ κύριο Φόξ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κασίνη για την έκθεση. Τα μέλη της ΑΦΚΟ και η Επιτροπή εργάστηκαν ώστε να μπορέσουν ε, να εργαστούν επικοδομητικά ώστε να υπάρχει σε όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία περισσότερη διαφάνεια. Κυρία Πρόεδρε, καλό που είστε εσεί, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την δουλειά που επιτελέσετε για τι διαπραγματεύσει μεταξύ τη Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση αυτή είναι μια σωστή έκθεση και χρήσιμη και νομίζω ότι θα είναι θετική και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει στα πλαίσια της κοινοτική νομοθεσίας και στην ε, ισόρροπη σχέση μεταξύ των ε, αυτών που κάνουν το λόμπι και της τοπικής αυτοκίνησης. Πολλά θα πρέπει να γίνουν όμως ακόμη και ελπίζω ότι αυτό το Μητρό, εάν ε, είναι επιτυχές, θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε ένα υποχρεωτικό Μητρό για τους λόμπις. Συμφωνώ με τον κύριο Νταφ ότι θα πρέπει οι εισηγητές να καταγράφουν τα ονόματα των εκπροσώπων των λόγων με τους οποίους ήρθαν σε επαφή όταν κάνουν καμιά έκθεση. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε διαφάνεια και σε ανοίγμα κάτι το οποίο ζητούν και οι ψηφοφόρες. Επιτρέπεστε μου επίσης να πω ότι το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι δεν έχουμε ε, λείπει ένα θεσμικό όργανο. Δεν έχει υπογράψει ακόμη ε, τίποτε το Συμβούλιο και η περαιτέρω συνεργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι σωστό και διαφανές. Ο κύριος Χέφνερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πολιτική χρειάζεται εμπιστοσύνη. Τα μέλη αυτού του κοινοβουλίου είναι ερετά σε ε, μυστική ψηφοφορία από τους συμπολίτε μας και αυτοί αναμένουν σε όλες τις ομιλίες μας και στις αποφάσεις μας να έχουμε στο νου μας το κοινό καλό, το ε, καλό των πολιτών και όχι τα συμφέροντα τρίτων εταιριών ε, ή άλλων. Ξέρουμε επίσης και το γνωρίζουν όλοι ότι γύρω μας υπάρχουν πάνω από 10.000 ε, επαγγελματίες ε, λομπίστες οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή να επηρεάσουν μέλη των επιτροπών. Πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό. Ζούμε σε μία ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία, αλλά πρέπει να μπορούμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε την ε, ανεξαρτησία μας. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη πάντοτε. Ορισμένοι ε, ε, βουλευτές παραβίασαν τον κανόνα αυτό και γι' αυτό τώρα κοιτάμε πώς θα βελτιώσουμε την ε, κατάσταση αυτή εξού και εκπονήσαμε αυτό το μητρό διαφανείας από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό όπως είπα θα προτιμούσα από την αρχή να έχει συμμετάσχει και το Συμβούλιο. Η πράσινη ήταν πάντοτε υπέρ αυτού του εγχειρήματο. Χαιρόμαστε που παρόλο που δεν μας ικανοποιούν όλοι. Θα θέλαμε να είναι δεσμευτικό, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και προς τα έξω. Δηλαδή το να πιει κανείς ένα κρασάκι σε ένα εστιατόριο στο Βέλγιο. Και αυτό όχι μόνο εις, ε, σε ορισμένα θεσμικά ε, όργανα, αλλά και στο Συμβούλιο και γι' αυτό τα μικρά εγχειρήματα χρειάζονται μικρά προγράμματα και τα μεγάλα πολύ πιο μεγαλεπίβολα κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία κοινή τελική γραμματεία αλλά αυτά είναι όλα καλά για τη διαφάνεια στην Ευρώπη και ευχαριστώ όλους αυτούς που συνέβαλαν στην υλοποίησή του. Ευχαριστώ κύριο Σόντεγκάρτα από την ε, Νοτική Αριστερά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Χρειάζεται πλέον περισσότερη διαφάνεια και ένα υποχρεωτικό μητρό ε, όπου να αναγράφονται όλοι εκείνοι που προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας όμως και όπως έδειξαν ε, διεφθαρμένοι ευρωπουλευτές θα πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε το ίδιο μας το σπίτι πριν μιλάμε για οτιδήποτε παραπάνω. Δεν είναι δυνατό ε, εκλεγμένοι ευρωβουλευτές ε, από τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν και κάποια πάρεργα και μάλιστα αμοιβόμενα και παράλληλες δραστηριότητες. Χρειάζονται σαφείς κανόνες προστασίας εκείνων που αποκαλύπτουν τέτοιες καταστάσεις για να μην τιμωρούνται εκείνοι αλλά οι πραγματικοί υπέτη. Χαιρόμαστε που η έκθεση τη έκτακτη Επιτροπή ε, τώρα είναι επιτάπητο και ε, προσβλέπουμε σύντομα να εγκριθεί η συμφωνία που μας απασχολεί σήμερα για την αλλαγή του κανονισμού. Ευχαριστώ. Μια γαλάζια κάρτα θα δεχτείτε από τον κύριο Χαντ Πέτερ. Μάρτιν, παρακαλώ, κύριε Σόνταγκάρτ. Έχετε το λόγο, κύριε Μάρτιν. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να ρωτήσω τι ε, σκέφτεστε για την πρόταση του νομοθετικού αποτυπώματος. Και γιατί δεν θα πρέπει να είναι το μητρό ε, υποχρεωτικό και δεσμευτικό, τα ε, θυράκια παραμένουν. Ε, Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να τονίσω και πάλι κάτι που είχα πει στην αρχή. Θα πρέπει ακόμα να επιτύχουμε πολλά. Δεν θεωρούμε ότι έχει λήξει η υπόθεση. Ε, παραμένουν ακόμα πάρα πολλά να γίνουν και ε, οπωσδήποτε αυτό το θέμα του δεσμευτικού χαρακτήρα του υποχρεωτικού μητρώου ε, είναι αποφασιστική σημασία. Σε ό,τι αφορά το, νομοθετικό, όπως είπατε, αποτύπωμα, το ηλεκτρονικό, καλό μου φαίνεται και θεωρώ θα πρέπει να μετεξελιχθεί. Και, αλλά όλα φυσικά για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι δεσμευτικά ή υποχρεωτικά. Ένα πρώτο βήμα έχει γίνει και ελπίζουμε όταν έρθει η έκθεση της έκταξης επιτροπής και την επεξεργαστούμε να προχωρήσουμε. Εξάλλου σε δύο χρόνια ε, επίκειται θέωρηση. Θα πρέπει να φτάσουμε οπωσδήποτε στο στόχο μας. Ευχαριστώ. Από την ομάδα του το λόγο έχει τώρα ο κύριος Άγνου για ένα λεπτό. Θέλουμε δηλαδή ένα μητρό διαφάνεια. Καθόλου δεν μας α, εκπλήσει, γιατί φαίνεται ότι μια βρετανική εφημερίδα με πολύ εύκολα αποκάλυψε πώς ενδίδουν στον πειρασμό του χρήματος ε, πολλοί ευρωβουλευτές. Βέβαια, ε, μερικοί διέριξαν τα ημάτια τους που ανακαλύφθηκε αυτό το λόμπι ε, ε, και ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν κάνουμε τίποτα γιατί σχεδόν τίποτα δεν θα αλλάξει με το Μητρό Διαφάνειας, θα παίρναν πάντα οι ομάδες πίεσης. Είχαμε ένα σύστημα καταχώρησης, αλλά ήταν αναποτελεσματικό. Τώρα υποτίθεται ότι θα λάμψει λίγο φως, θα χυθεί λίγο φως, αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα αποτελματωθεί η κατάσταση και δεν θα αλλάξουν και πολλά. Τελικά οι έντιμοι θα υποστούν το άχθος της γραφειοκρατίας, ενώ οι άτιμοι θα βρουν κάποιο παραθυράκι για να διεισδύσουν. Φαίνεται ότι δεν θα πατάξουμε τα ανενδίαστα λόμπι, γιατί μονίμως υπάρχουν όροι να προσπαθούν να κατασπαράξουν άλλη γαλάζια κάρτα σηκώθηκε από τον κύριο Χέφνερ. Θέλετε να απαντήσετε, είστε... Δέχεστε να απαντήσετε στην ερώτηση, αν την καταλάβω. Αγαπητέ συνάδελφε, είμαι πολύ υπέρμαχος μιας αξιοπρεπούς ανταλλαγής ε, επιχειρημάτων και διαξυφισμό σε μια ε, αντιπαράθεση. Αλλά ε, εκνευρίζομαι όταν ακούγονται λάθη. Είπατε ότι το συζητάει το κοινοβούλιο αυτό μόνο επειδή πρόσφατα κάποιοι Άγγλοι δημοσιογράφοι κίνησαν το θέμα. Μπορείτε σας παρακαλώ να εξηγήσετε στην κοινή γνώμη ότι δεν αρχίσαμε τώρα εδώ, ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια για το Μητρό Διαφάνειας και μάλιστα έχει ολοκληρωθεί πριν συμβεί η ιστορία την οποία έχετε υπόψη σας. τώρα, αν ήταν αφορμή ή ο καταλήτης, ε, εγώ δεν θα δεν πιστεύω ότι καν δικαιολογεί την παρουσία των Βρετανών εδώ, γιατί δεν είμαστε υπέρ τη καθοδήγησή μα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω άλλο να... θέλω άλλους να ελέγχουν τα πράγματά μας. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε τμήμα αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλτσερ. Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ε, ε, υποφέρει από ένα μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας και το κοινοβούλιο αλλά και κάτι άλλο που δεν ε, αρέσει το κοινοβούλιο να τα ακούει επιτέλους ε, ε, κατάφερε να συμφωνήσει και μετά από αυτά τα τελευταία με τους δημοσιογράφους, αλλά τελικά είναι ξεδοντιασμένη αυτή η προσπάθεια. Είναι υποκριτικό και μόνο για τα μάτια εφόσον δεν είναι δεσμευτική η καταχώρηση. Ε, αφήστε δε που το Συμβούλιο απέχει, δηλαδή ο άλλος σημαντικός νομοθέτης. Και ακόμα και αν συμμετείχε θα ήταν τεράστια ακόμα τα παραθυράκια. Εκατοντάδες υποτίθεται Υπάρχουν ε, εμπειρογνώμονες και ε, διάφοροι κύκλοι που συνεχίζουν να συνεδριάζουν και κλεισμένο το θυρών και αυτό είναι επτασφράγιστο μυστικό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να καταγράφονται ε, μόνο οι οικονομικοί όμιλοι αλλά και άλλοι εκπρόσωποι συμφερόντων που πληρώνονται και αμείβονται όπως είναι τα συνδικάτα και τα επιμελητήρια. Έχει δικαίωμα ο πολίτη στη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιαννάκου παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Καζίνη ε, για την έκθεσή του η οποία είναι πολύ σωστή. Βέβαια η υπόθεση της διαφάνειας επαφίεται κύριε Πρόεδρε στην αξιοπρέπεια των βουλευτών δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά όσο περισσότερα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα παίρνουμε, τόσο προωθούμε ουσιαστικότερα τη διαφάνεια και τη λειτουργική σχέση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις ομάδες συμφερόντων. Το νέο Μητρό, όπως προτείνεται, διασφαλίζει διαφάνεια για το ευρυφάσμα επαφών των θεσμικών οργάνων και συγκεκριμένα συγκεντρώνει σε χωριστά κεφάλαια εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους των δημοσίων αρχών και με αυτόν τον τρόπο διακρίνει τους διαφορετικούς ρόλους των ομάδων συμφερόντων και των επισήμων συνομιλητών των θεσμικών οργάνων. η πρόσκληση για καταχώρηση στο μητρό διασφαλίζει την ίδια την ταυτότητα των ομάδων συμφερόντων και των λομπίστ, καθώς τους αναγνωρίζει αυτοτέλεια και τους θέτει σε επίπεδο άμεσης και απευθείας συνομιλίας με τα θεσμικά όργανα τη Ένωση μετά την κύρωση της συνθήκης της λισαβόνας οι εξουσίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου είναι ενισχυμένες και προσελκύουν κατά συνέπεια όλο και μεγαλύτερο ε, αριθμό εκπροσώπων συμφερόντων που αναζητούν παρεμβάσεις. εν κατακλείδη κύριε πρόεδρε το μητρό διαφάνειας υπηρετεί κατά κύριο λόγο τη διαφάνεια και τη δημοκρατική και πλουραλιστική διάδραση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους στους εντολείς των βουλευτών που είναι οι πολίτες ο λαός και τα θεσμικά όργανα της ένωσης. εξυπακούεται βέβαια ότι σε ένα τέτοιο μητρό διαφάνειας υποχρεωτικά πρέπει να έχουν θέση όλα τα mm. όργανα και τα στελέχη της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Κασίνη για τις ε, εκθέσεις του για τα Μητρώα Διαφάνειας. Διανύουμε μία κρίση τεραστίων διαστάσεων που σοβεί εδώ και καιρό και μάλιστα απειλεί να παραμείνει ακόμη περισσότερο καιρό. Και σε τέτοιου είδου κρίσει ε, ε, όχι μόνο το βιωτικό επίπεδο πλήττεται των κατοίκων, των πολιτών της Ένωσης, αλλά και το μέλλον τους, οι ελπίδες τους. Θα πρέπει λοιπόν με τις πολιτικές μας και με τα θετικά αποτελέσματα που θα έχουν να συμβάλλουμε στη νομοποίηση και στην σαφή τήρηση των αρχών της αυστηρότητας, της λιτότητας, της διαφάνειας, της εντιμότητας και της προσέγγισης στους πολίτες. Και αυτό το Μητρό είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας. Ένα βήμα μόνο όμως είναι. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που τόνισαν ότι θα πρέπει το Μητρό να γίνει υποχρεωτικό, να συμπεριληφθεί και στο Συμβούλιο και να περιλαμβάνει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που εντοπίζονται ατασταλίες ή παράτυπες συμπεριφορές. Η κυρία Τάιν τώρα, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο όταν θα ψηφίσουμε για το Μητρό διαφάνεια. αυτό θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και η απόλυτη και τελική λύση. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι ε, το Μητρό των Ομάδων Πίεσης που υπάρχει το 1996 το μετονομάζουμε σε Μητρό διαφάνεια. Γιατί σκεπτόμενοι το πόσοι πρέπει να καταγραφούν για να πάρουν ε, την ε, κάρτα εισόδου σε όλους τους οργανισμούς που έχουμε εδώ, ε, σκεπτόμενοι όλα αυτά, κατανοώ βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει ένα μητρό. Εκείνο όμως που δεν κατανοώ είναι ότι ε, ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου που εξορισμού δεν πρέπει να τοποθετείται πολιτικά και δεν τοποθετείται θα πρέπει να καταγραφεί. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μορφή διαφάνειας, σε τελική ανάλυση ο κάθε ευρωβουλευτής έχει τη δική του την πηξίδα για να τον οδηγήσει τι είναι σωστό και τι όχι. Μόνος το αποφασίζει ποιον θα συναντήσει ε, ποιον ε, θα, ε, με ποιον θα διαβουλευτεί, γιατί στη τελική ανάλυση πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να μας πλησιάσουν. Κύριος Μάρτιν, παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό με την εσωτερική πηξίδα είναι ένα μεγάλο θέμα. Βεβαίω και πρόκειται για την ανεξαρτησία των ευρωβουλευτών και η πίεση των πολιτικών ομάδων δημιουργεί πρόβλημα. Οποτεδήποτε καταβάλλονται προσπάθειες να ε, μετατρέψει κανείς την άποψη ενός ανθρώπου. Αυτό κυρίως όταν πρόκειται για ε, αθέμητες πρακτικές. Στην, ε, στις είναι 2.000 τόσοι ε, που εκπροσωπούν ομάδες πίεσης. Εκείνο που είναι γεγονός ε, και θέλω να το πω είναι ότι εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Με αυτό λοιπόν το, διαφάνιο το μητρό διαφάνειας κάνουμε ένα σωστό βήμα αλλά κατ' ουσίαν θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Ουάσιγκτον. Γιατί εκεί υπάρχει ένα μητρό που λειτουργεί πολύ καιρό και είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε εμεί εδώ. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε προφανώ ε, ένα βήμα προ τη νομοθετική κατεύθυνση, αλλά ένα μεγαλύτερο βήμα. Μόνοι μα θα αποφασίσουμε με ποιου ερχόμαστε σε επαφή, ε, τι θα συζητάμε μαζί του ε, και εγώ στη δική μου την ιστοσελίδα ίντερνετ έχω ένα link όπου δείχνει ότι ε, ανεξάρτητα με το αν εργάζομαι σε μια νομοθετική πρωτοβουλία ή όχι, φαίνεται με ποιου εκπροσώπου ομάδων πίεση έχω έρθει σε επαφή και με ποιου όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προετοιμάζουμε τους κανόνες που θα ισχύουν. Δημιουργείται η εντύπωση ότι η... Ε, διαφθορά και τα προνόμια υφίστανται, ενώ στην, ε, επί της ουσίας πρόκειται για ανθρώπους με ειδική τεχνογνωσία που θέλουν να μας ενημερώσουν και οι οποίοι ε, θέλουν να τοποθετηθούν πάνω στα νομοθετήματα που θεσπίζουμε. Ας πούμε, για την προστασία των δεδομένων. Ήρθαν πολλοί και με βρήκαν ε, για να τοποθετηθούν και αυτό με εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πω το εξή. Αν εγώ ήμουν αναγκασμένος να καταγράφω ε, εκείνους που έρχονται να με βρουν, ε, αυτό ίσως να ήταν σωστό, γιατί με τον τρόπο αυτό θα είχαμε πλήρη διαφάνεια. Εγώ, κοιτάξτε, καταγράφω εκείνους που έρχονται σε μένα, αλλά και πολλούς άλλους για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια Σας ευχαριστώ πολύ. Ο αντιπρόεδρο και αντιπρόεδρο τη ομάδα εργασία, ο κ. Λαμπρινίδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ συχνά λέμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε αγνοούν τι ε, τεράστιε νομοθετικέ αρμοδιότητε που προσθέθηκαν μετά τη Λισαβόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά είναι ατυχέ. Πάντω, οι λόμπι αυτοί που κάνουν ε, του λομπίστε, όπω πρόσφατα, φαίνεται ότι ξέρουν πολύ καλά τις νομοθετικέ εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί συνομοθετούμε σχεδόν σε όλα τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα είμαστε το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρόλο που αυτό ισχύει και θα είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια, ένα από τα πιο διαφανή θεσμικά όργανα, πιστεύω ότι μαζί με την αύξηση των εξουσιών έχουμε και περισσότερη ευθύνη και μεγαλύτερη υπευθυνότητα και συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Κασίνη. Δεν είναι κακή αυτή η έκθεση. Αλλά θα πρέπει να υποχρεούνται τα λόμπι ομάδες πίεσης να αναφέρουν, να εγγράφονται με ονόματα και τα συμφέροντά τους στο Μητρό. Και ελπίζω να μας μιμηθούν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα με αυτή την καταγραφή των λόμπι. Όπως είπατε είμαι και αντιπρόεδρος της σχετικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε για τι συζητήσει αυτή τη ομάδα. Σα διαβεβαιώ πάντω ότι θα φροντίσουμε οι δαντολογικοί κανόνε και οι κώδικε συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι από του πιο διαφανεί και θα κάνουν τους ε, πολίτες μας ε, και εμάς περήφανους ε, για το ότι είμαστε μέλη αυτού του καταπληκτικού θεσμικού οργάνου. Και τώρα η κυρία Φλασίκοβα Πένοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Μπορεί να βελτιώνει την κατάσταση το Μητρό, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, απέχουμε πόρο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και οι εκπρόσωποι των ομάδων πίεση ξέρουν ότι εάν δεν εγγραφούν σε αυτό το Μητρό δεν θα έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο. Και θα του γνωρίζουμε και εμεί καλύτερα και τα ονόματά του ε, και όσοι δεν ε, συμμορφώνονται προς ε, τις διατάξεις θα υφίστανται και συγκεκριμένες κυρώσεις. Το θέμα δεν ξέρω αν ακούν όλα αυτά. Η καταχώρηση στο κοινοβούλιο ουσιαστικά είναι υποχρεωτική για να έχουν πρόσβαση, επαναλαμβάνω, στο, κοινοβούλιο, στο κτίριο του κοινοβουλίου. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να υποχρεώνονται και de jure, όχι μόνο de facto. Μέχρι τέλους της παρούς θα πρέπει το Κοινοβούλιο να το έχει αποφασίσει αυτό. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε και πιο ακριβή ε, στοιχεία. Και... Ως προς το κόστος ε, και τα οικονομικά που συνδέονται με τις δραστηριότητες των ομάδων λόμπι. Σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν αυτά σε ό,τι αφορά τώρα τον κώδικα διοντολογίας, παρακαλώ να μην συγχαίρετε με το Μητρό Διαφάνεια. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν πέσει θύματα ε, κάποιου σκανδάλου πρόσφατα και θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό το θέμα, αλλά ξεχωριστά να μην το συγχαίουμε. Η κυρία Ολτσκόκ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν. Δεν πειράζει να τα επαναλάβω κι εγώ. Ε, συμφωνήσαμε για ένα μητρό ε, που θα καταγράφονται τα λόμπι. Πολλοί από εμά έχουμε αγωνιστεί πολύ καιρό. Ε, Παρ' όλα αυτά παραμένει μετριοπαθής και προσεκτική η πρόταση. Εν είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για ε, μια πολύ ε, μεγάλη προσπάθεια διαφάνειας σωστά και ωραία και αυτά που είπε και ο Επίτροπο Εύκοβη και το Συμβούλιο. Η διαφάνεια είναι πραγματικά σημαντική για να περιοριστούν οι κίνδυνοι ε, καταχρήσεων. Και επίσης να αυξηθεί η εμπιστοσύνη για μα, τους ευρωβουλευτέ και την πολιτική γενικότερα. Θα πρέπει όμως να ε, συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα σε ένα τέτοιο μητρό διαφάνεια. και να είναι υποχρεωτικό και να συμπληρώνεται όπως συμβαίνει άλλωστε και στις σκανδιναβικές χώρες. Με προστασία εκείνων που καταδεικνύουν τα κακό σκήμενα και τα αποκαλύπτουν, του λεγόμενου whistleblowers. Παίρνουμε στη διαδικασία CatchDI τώρα, λέει ο πρόεδρο. Ο κ. Μικολάσικ είναι πρόεδρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σεύκοβιτς, κύριε ε, Υπουργέ Γκέρι, η δημιουργία του Μητρώου Διαφάνειας για τις ομάδες πίεσης που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί. Πραγματικά χρειάζεται ε, να έχουμε σαφείς κανόνες και αυστηρούς κανόνες και αυτό αποτελεί εγγύηση της ε, σωστής και δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Βεβαίως θα πρέπει και οι ευρωβουλευτές να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την εντολή που τους έχει δοθεί και να έχουν τη δυνατότητα να συναντούν και πολίτες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ε, θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ σαφείς κανόνες, επαναλαμβάνω, μια ειλικρινής και ε, διαφανή συζήτηση με εκείνους που συμμετέχουν και θέλουν να επηρεάσουν τη δομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ. Λαμβάνω το λόγο ως εισηγητής ε, της πρόσβασης του κοινού ε, στα έγγραφα του κανονισμού 1049 και νομίζω ότι το πνεύμα της διαφάνειας ε, ε, διέπει και αυτόν τον κανονισμό του 2001 και είναι το βήμα προς σωστή κατεύθυνση γιατί η διαφάνεια βρίσκεται στην καρδιά της διαδικασίας λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ε, ποιοι επηρεάζουν και μερικές φορές ε, αδίκως ε, τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και την έκβασή της. Θα πρέπει όμως να επιτείνουμε το έργο μας ώστε η διαφάνεια και η ακαιρεότητα του έργου των ομάδων πίεσης να υπόκειται σε υψηλέ προδιαγραφέ. Και θέλουμε το νέο Μητρό Διαφάνεια ε, να ισχύσει το συντομότερο δυνατό. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει όλα τα πρόσωπα και όλε οι οργανώσει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του Μητρώου να παρέχουν ακριβεί και ενημερωμένε πληροφορίε για να βλέπουμε ποιο επηρεάζει τι. Και τέλο, όπω είπε ο Γιάννα Μίτεμαερ από την Διεθνή Διαφάνεια, το νέο Μητρό θα αποτελέσει λιδία λίθο για τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων σε ό,τι αφορά την ε, πίεση προς, μια μεγαλύτερη, προς ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Νομίζω ότι ε, το σαφές και το λακωνικό. Η κυρία Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο, αιώνας, ε, ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας του διαδικτύου, της Wikileaks, του διοργανικού ανοίγματο, τη συμμετοχή του πολίτη και τη διαφάνεια. Θα πρέπει όμω να ευαισθητοποιηθούμε και να συγκροτήσουμε σωστά τι αποφάσει μα. Να συνεργαστούμε. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε δραστήριοι. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να μα ασκούν πιέσει οι λόμπι ομάδε πίεση. Θα πρέπει εμεί να πλησιάσουμε του Ευρωπαίου πολίτε, να ακούσουμε τη γνώμη του. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι αποτελεσματικό το Μητρό διαφάνεια και ε, το ψηφιακό αποτύπωμα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε έτσι και τις εκθέσεις μας και να καταμετρήσουμε τα αποτελέσματά τους, γιατί έτσι θα βαδίσουμε προς ένα σύγχρονο κοινοβουλευτισμό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε όλους τους συνεργάτες μας και αυτός είναι ο σωστός τρόπος ε, εργασίας για να διαχωριστούμε από τις ανεύθυνες συμπεριφορέ που μερικέ φορές παρατηρήσαμε στο παρελθόν. Η ε, κυρία Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι για το κείμενο που με ιδιαίτερη χαρά θα υπερψηφίσω αύριο. Και μάλιστα το πρόσφατο σκάνδαλο ήταν μια απόπειρα διαφθοράς και τίποτα παραπάνω. Σοβαρή μεν, αλλά αυτά τα πρόσφατα ε, γεγονότα δείχνουν ε, είναι πολύ μεταγενέστερα από τη δική μας προεργασία και τη δική μας προσπάθεια διαφάνειας που είναι πολύ παλαιότερη. Και το τελευταίο σκάνδαλο είναι μεμονωμένο. Σίγουρα οι προσπάθειες ε, ομάδων πίεσης είναι σημαντικοί και θα κάνουν ε, προσπάθειες να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό και το Μητρό είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Συνέβαλα στην κατάρτισή του και χαίρομαι για το αποτέλεσμα αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλα βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει το Μητρό αυτό να μετατραπεί σε ένα δυναμικό και όχι στατικό ε, και ακίνητο όργανο, γιατί η κατάσταση εξελίσσεται. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματικότητά του και να βλέπουμε ποιο λόμπι για πόσα χρήματα και με ποιο τρόπο προσπαθεί να επηρεάσει τα πράγματα. Και συμφωνώ και με το νομοθετικό αποτύπωμα, θα έλεγα οικολογικό κατά, κατά λάθος. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι λομπίστες, πόσους ε, συνάντησαν, ποιος είπε τι, ποιος επηρέασε ποιον. Θα πρέπει επίση ε, να δώσουμε εξηγήσει για το πώ λειτουργεί η κατάσταση, γιατί αυτό χρειάζονται οι πολίτε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Μητρό και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καταλαβαίνουν πώ ε, λειτουργεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και θα υπερψηφίσω αύριο. Ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ε, οι ομάδες πίσης είναι πολύ σημαντικές για τη συμμετοχή των πολιτών και γι' αυτό είναι εξίσου σημαντικό να παρεμποδίζουμε καταχρήσεις. Χρειαζόμαστε επιγόντω μητρό για όλου του θεσμού. Όχι μόνο για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και για το Συμβούλιο. Γιατί εκεί λαμβάνονται επί τη ουσία οι αποφάσει. Και κάτι άλλο. Η καταγραφή πρέπει να είναι δεσμευτική, όχι μόνο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο, γιατί οι εκπρόσωποι των ομάδων πίεση ε, έρχονται σε επαφή με του ευρωβουλευτέ, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε δεξιώσει και σε γυμναστήρια. Και να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά τη διαφάνεια των κομμάτων, ακόμα και αν είναι πρόσωπο τα κόμματα ε, και ακόμα και αν εμφανίζονται ως ε, επιχειρήσεις ή ως ε, τα καθαρά χέρια της Ευρώπης και αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς, να καταγράφονται, θα πρέπει επίσης να παραθέτουν τα στοιχεία για τις πραγματικές δαπάνες που, ε, ε, ε, τις οποίες πράττουν, τις οποίες εμφανίζουν στη διάρκεια των προκλογικών εκστρατιών. Και θα πρέπει και σε αυτό το θέμα λοιπόν να επικρατεί διαφάνεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτό που είπαν οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ, ότι το Μητρό αυτό αποτελεί μια πρόοδο ό,τι αφορά την εξασφάλιση διαφάνεια τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, όμω, αυτό το. Ε, αυτό το βήμα είναι ένα και μόνο βήμα και θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες λύσεις και άλλα βήματα. Κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό είναι η απάντηση στην ερώτηση τι δίνεται ο Ευρωβουλευτής. Ο Ευρωβουλευτής εργάζεται μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι το επάγγελμά του, ή εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει και άλλε δραστηριότητε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτέ οι άλλε δραστηριότητε θα πρέπει να ερμηνευτούν πολύ συσταλτικά και να περιορίζονται σε δημοσιεύσεις ή σε επιστημονική εργασία. Οποιαδήποτε άλλες δραστηριότητες όπως συμβάσεις κτλ. θα γύρουν αμφιβολίες και υπόνοιες. Και ο τελευταίος ομιλητής, η κυρία Εκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει πλέον ε, μεγαλύτερες αρμοδιότητες, εξουσίες αλλά και ευθύνη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς νομοθετούμε για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Συχνά ε, συνδέεται και μεγάλο οικονομικό κόστος με αυτά. Το Μητρό Διαφάνειας λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι πολύτιμο και ελπίζω να προχωρήσουμε και να ε, προστατεύουμε και εκείνους που αποκαλύπτουν ε, τα κακό να δίνουν πληροφορίες και ε, θέλω να είναι υποχρεωτικό το Μητρό όχι εθελοντικό, όχι προαιρετικό για το πόθεν για τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, αλλά και τις παράλληλες δραστηριότητες ε, που επιτρέπονται από πλευράς ε, ηθικής και δεντολογικής. Εν πάση είναι καλό βήμα, αλλά χρειάζονται πολλά βήματα ακόμα που πρέπει να γίνουν για μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δημοκρατία και περισσότερο η εμπιστοσύνη. Ο κύριος Σέφροβιτς έχει το λόγο για να συνοψίσει, να ολοκληρώσει, να κλείσει και να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις των μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι ο υπουργό τα είπε καλύτερα από όλου. Το Μητρό διαφάνεια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει περήφανος. Με ξέρετε τι Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά δεν γνωρίζω κανένα άλλο όργανο που να υπάρχει ένα τέτοιο μητρό και να λειτουργεί. Με ξέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Μιλώ και για τις πρωτεύουσε της ίδιας των κρατών μελών, έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα αντίστοιχα κοινοβούλια. Ε, πολύ με ρώτησαν και ο κύριος Γκρότε και ο κύριος ε, Χέφνερ για το κατά πόσο θα είναι υποχρεωτικό το Μητρό. Το συζητήσαμε διαμακρόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σήμερα δεν βλέπουμε την νομική βάση εκείνη που να μας ε, ε, επιτρέπει να υποχρεώνουμε εταιρείε, πολίτες ή εκπροσώπους γενικότερα να καταγράφονται για να ασκούν το επάγγελμά τους. Εμείς δεν έχουμε νομική βάση για να αρνηθούμε σε κάποιον συνεργασία μαζί του. Γι' αυτό Καλύτερα να προχωρήσουμε στη θετική ενθάρρυνση εταιριών, οργανώσεων και λόμπι να καταχωρηθούν εθελοντικά. Με την πυθό μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Συμφωνία με το Κοινοβούλιο μπορούμε να μετατρέψουμε το σύστημα αυτό σιγά σιγά σε υποχρεωτικό. Και ε, αν δεν συνεργαστούμε δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Αντίθετα, αν συνεργαστούμε και με το Συμβούλιο, θα αυξηθεί η πίεση σιγά σιγά και θα δούμε πώ θα λειτουργήσει το σύστημα την επόμενη διετία, έτσι ώστε να έχουμε και επιπλέον εμπειρία να κάνουμε την αναθεώρηση με ε, στοιχεία με μεγάλη ποιότητα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα, στην εξακρίβωση των οικονομικών συμφερόντων και οικονομικών δραστηριοτήτων, ε, τον λόμπι. Πρέπει να σας πω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους ε, των όσων ήδη είναι γεγραμμένοι στο Μητρό και πιστεύω ότι θα έχουμε και κοινό το ε, Μητρό θα γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Και να είναι βέβαιοι όλοι οι εγγεγραμμένοι ότι αν υπάρχει κάτι το αξιόμεμπτο θα το βρούμε, ε, θα το αναλύσουμε, θα τους τιμωρήσουμε και θα δημοσιοποιήσουμε και τα ονόματά τους. Θα επανέλθω συνέχεια σε αυτό γιατί πολλοί αναφέρθηκαν ε, και στα τρία θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να συμμετέχουν και τα τρία θεσμικά όργανα στο Μητρό. Μετά από ε, ε, την έναρξη των διαπραγματεύσεων επί Ουγγρικής Προεδρίας νομίζω δεν θα αφιστούμε χρόνο και πάρα πολύ ε, γρήγορα θα προχωρήσουν οι εργασίες, ε, οι συνεννοήσεις για να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν και τα τρία θεσμικά όργανα πάντα με στόχο την αύξηση της διαφάνειας ε, στη παρασκευαστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τελευταίο που πάλι αναφέραν πολλοί βουλευτές και ο κύριος Καζίνη ο ίδιος. Το Μητρό Διαφάνειας Βεβαίω, ούτε πανάκια είναι ούτε μαγική λύση για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Ε, ξέρουμε ότι ε, οι αρχές, οι αξίες, ε, η ηθική και οι σαφείς κανόνες από κοινού θα πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μας. Πάντως οι κανόνες είναι δεδομένοι και εκείνοι που καταγράφονται είναι πρόθυμοι να τους ακολουθήσουν, ε, δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, συμφωνούν να προχωρήσουν έτσι και αυτό θα πρέπει να είναι ο γνώμονάς μας. Να συνεργαζόμαστε, να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες που έχουμε και να εμπιστευόμαστε τη μελλοντική μας επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυρία Γιώρη, εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Ως πολίτης κράτου κράτους θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή τη συζήτηση και μάλιστα όχι μόνο συζήτηση, αλλά και τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του Μητρώου Διαφάνειας. Είμαι πολίτης μιας χώρας που από το 2006 έχει νομοθεσία που διέπει το ζήτημα της δραστηριότητας των ομάδων πίεσης. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για μας. Και χαίρομαι που στη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας το Συμβούλιο είναι έτοιμο να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία και να συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην ε, πρόθεση αυτών των εργασιών για το Μητρό Διαφάνεια. Το Συμβούλιο είναι πια έτοιμο και ανοιχτό για διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η αγαστή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Και μάλιστα αυτή η βούληση του Συμβουλίου θα πρέπει να μεταφραστεί και σε μια πολιτική διακήρυξη τον Ιούλιο. και νομίζω ότι η διοργανική συμφωνία είναι το μόνο που μπορούν να δεχτούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτό θα σημάνει και την αισθητή πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το Συμβούλιο βέβαια δεν είναι ένα θεσμικό όργανο που βάλεται από τις ομάδες πίεσης, που κατακλείζεται από ομάδες πίεσης. Οι λομπίστες και οι ομάδες πίεσης πηγαίνουν περισσότερο στις κυβερνήσεις, στα κράτη-μέλη για να δώσουν την γνώμη τους. Το Συμβούλιο είναι λιγότερο εκτεθειμένο στις δραστηριότητες των ομάδων πίεσης. Πολύ λιγότερο σίγουρα από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως είμαι βεβαία ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και μετά τις διαπραγματεύσει θα καταφέρουμε να καταλήξουμε τον Ιούλιο στην πολιτική διακήρυξη. Και ο κύριος Κασίνη, ο εισηγητής μας, θα έχει το τελικό λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω μόνο κάποιες διευκρίνησεις και εγώ θέλω να επισημάνω κατηγορηματικά ότι πράγματι αυτή η συμφωνία ε, συμφωνήθηκε, συνήφθη λίγο πριν γίνει αυτό το σκάνδαλο με τους ε, Άγγλους δημοσιογράφους. Μην ξεχνάτε ότι οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ε, ε, μπέζουν όπως η Κοριέρα Ντελασέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα δηλαδή πολύ σωστά καταλαβαίνετε ότι φύγουμε το θέμα της έλλειψης εμπιστοσύνης από, ε, απέναντι στην Ευρώπη. Και αυτή η συμφωνία συνήφθη λίγο πριν γιατί από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο διερωτηθήκαμε κατά πόσο μπορούμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τη συμφωνία. Η συμφωνία όμω, όπω σα λέω, είχε ήδη συναυθεί προηγουμένω και αυτή είναι μια διευκρίνηση. Κατόπιν, το κατά πόσο είναι δεσμευτικό το Μητρό είναι δεσμευτικό. Όποιο ε, θέλει να αποκτήσει δικαιώματα του πρέπει να καταγραφεί στο Μητρό αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει περαιτέρω από αυτό ε, ε, υποχρεωτικό. Δηλαδή ότι πρέπει εκεί να καταγραφούν όλοι οι πολίτε τη Ευρώπη. Μα αυτό είναι αδύνατον. Αν κάποιο θέλει να ασκήσει πίεση, θα πρέπει πρέπει να καταγραφεί. Αυτό βέβαια είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τρίτη παρατήρηση οι μελλοντικέ τροποποίησει από την ομάδα εργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτήν την ομάδα εργασία να δώσουμε ω το δυνατόν περισσότερο λιγμών. Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο ε, να ε, επισημάνουμε το γεγονός αυτό στους ε, εκπροσώπους της ποιησης ε, κατά τη διάρκεια των επαφών. Θα πρέπει όμως το Μάντρα εργασίας να δώσουμε πλήρη ελευθερία για να καταθέσει τις απαραίτητες προτάσεις. Τελευταίο σημείο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και τον ε, Επίτροπο που πραγματικά συνέβαλε στο να συναυτεί αυτή η συμφωνία και στην εκπρόσωπο, στους εκπροσώπους της Ουγγρικής κυβέρνησης, συγκεκριμένα στην κυρία για τις διευκρινήσεις που μας έδεσε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο. Ας μην ξεχνάμε ότι και βεβαίως το Συμβούλιο είναι ε, ο δεύτερος θεσμός. Ε, γι' αυτό λοιπόν η επέκταση του Μητρώου σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε καλύτερα ότι η ε, αντιμετωπίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα εκτελεστικό οργανισμό. Θέλω όμως να κάνω και μία διευκρίνηση γιατί το Συμβούλιο των Υπουργών εκπροσωπεί τα κράτη και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μία άποψη η οποία θα είναι κοινή, θα τη συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε λοιπόν και θέλω να πω ότι ε, όσοι συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση έκλεισε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 12.30. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση για την ε, πυρηνική ασφάλεια 25 χρόνια μετά την καταστροφή στο Τσερνομπίλ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο